if you have questions afterwards, she's happy to take some. Please obviously say who you are and which media you represent. Commissioner. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ε, μόλις τέλειωσε μια διαδικασία πολύ δημοκρατική, αλλά και πολύ δύσκολη. Ε, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι μια διαδικασία τριών ωρών με ερωτήσεις από βουλευτές από όλα τα πολιτικά από όλες τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να ελπίζω ότι οι απαντήσεις μου ήταν οι σωστές και προσβλέπω σε έναν επικοδομητικό διάλογο με τους Ευρωβουλευτές. Γιατί Ιδιαίτερα σήμερα με την ε, συνθήκη της Λισαβόνας η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γίνεται ακόμη πιο απαραίτητη. Έχω, πιστεύω, την εμπειρία των τελευταίων δύο χρόνων στο ε, χαρτοφυλάκιο της υγείας το οποίο μου έδωσε την εμπειρία αυτή της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω θα μπορούσαν κάλλιστα να χτίσω πάνω σε αυτή την εμπειρία. Το καινούριο μου χαρτοφυλάκιο είναι χαρτοφυλάκιο πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα έλεγα ότι πολύ ενδιαφέρον ιδιαίτερα για την μικρή μου πατρίδα Κύπρο. Γιατί η Κύπρος δεν έχει ούτε μεταλλεύματα, ε, ούτε άλλες πηγές εσόδων εκτός από την φιλοξενία της και τον πολιτισμό της. Και πιστεύω ότι και η Κυπριακή Προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά τα θέματα γιατί είναι το δυνατό μας σημείο. Και έτσι είμαι πολύ ευτυχής που ανέλαβα αυτό το χαρτοφυλάκιο το οποίο πρέπει να σημειώσω είναι